Der Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Ξαναρχίζουμε τη συνεδρίαση λοιπόν, τελευταία πριν από τα Χριστούγεννα και τον καινούριο χρόνο. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να χαιρετήσω εδώ εκπροσώπους της Βάδης Βιτεμβέργης, της οργάνωσης για την υποστήριξη των θυμάτων πολέμων και ενόπλων αντιπαραθέσεων. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Okay, meine Ausführungen zum Protokoll erfolgen για τα πρακτικά. Θα κάνω παρατηρήσεις αργότερα. Στη συνέχεια έχουμε συζήτηση για, τα, για τις παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και έχουμε πρώτα το ζήτημα της Μαλαισίας. Η κυρία Βάιλερ